Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi ritengo opportuno iniziare, dare inizio ai lavori. Καλησπέρα. Ε, έχουμε καθυστερήσει λίγο. Νομίζω ότι καλό θα είναι να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους, ε, τα μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα τους ε, τρεις υποψήφιους. Πρώτο, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι έγκριση του σχεδίου ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, θεωρείται εγκεκριμένη η ημερήσια διάταξη. Να αναφερθώ στην ε, σημερινή διαδικασία. Η σημερινή συνεδρίαση είναι ανοιχτή σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τον ε, κανόνα υπαριθμών 204. Ε, η, ε, η Επιτροπή Αναφορών έχει έξι υποψήφιους για τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Μόνο τρεις υποψηφιώτες όμως γίνονται παραδεκτές σύμφωνα με τους κανόνες, με τι προποθέσει που αναφέρονται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε και σήμερα θα ακούσουμε τους ε, τρεις υποψήφιους με αλφαβητική σειρά, δηλαδή πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Βιτόριο Μπότολη, κατόπιν τον κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο και τέλος ε, τον κύριο Πιέρ Ιβ Μονέτ. Κάθε υποψήφιος έχει στη διάθεσή του μία ώρα. Μπορεί να παρουσιάσει καταρχήν την υποψηφιότητά του και κατόπιν να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών. Στο πρώτο τέταρτο θα ακούσουμε την παρουσίαση των υποψηφίων και μετά θα έχουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Και στο τέλος θα έχουμε και, μία, ε, και ένα τέταρτο για τη διαδικασία Catch the Στην ιστοσελίδα μας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών υπάρχουν όλες οι πληροφορίες σε σχέση με, τις, ε, με τη διαδικασία, οι, οι υποψήφοι που έγιναν δεκτοί και εκείνοι που δεν έγιναν δεκτοί. Επίσης έχουν εγγραφεί οι γραπτές ερωτήσεις και οι απαντήσεις των ιδίων. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα με αυτή την ακρόαση αλλά ήδη διαθέτουμε πληροφορίες τις οποίες λάβαμε από αυτή την προκαταρκτική διαδικασία από τους μεμονωμένους υποψηφίους. Στο τέλος της σημερινής ακρόασης, των σημερινών ακροάσεων μάλλον, η Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει και θα στείλει τη γνωμοδότηση στον πρόεδρο της, ε, του Κοινοβουλίου για να δούμε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας και η τελική εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αν δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ε, άρχεται λοιπόν η ακρόαση και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μπότολη να λάβει το λόγο. Non c'è. <laughs> sì, Θα, θα φτάνει τώρα, θα φτάνει τώρα. Μόλι φτάνει. Benvenuto. Allora, gli diamo qualche minuto per... Ας του δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα για να καθίσει. Και επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Μπότολη θα πρέπει να αρχίσει με μία παρουσίαση 15 λεπτών για να μας μιλήσει για τη δική του υποψηφιότητα και μετά θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής. Honorable President, honorable members of Committee of Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία μετά τον πρώτο γύρο επιλογής να εμφανιστώ εδώ. Η εισαγωγή μου θα είναι σκόπιμα σύντομη. Από την πείρα μου έμαθα ότι η συζήτηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αναπτύξω τα θέματα που θα επιλέξετε εσείς για να αξιολογήσετε καλύτερα το πρόσωπο που βρίσκεται μπροστά σας. Και είναι ο καλύτερος τρόπος για να αφήσουμε χώρο για οποιοδήποτε άλλο θέμα πιστεύετε ότι αξίζει την προσοχή σας. Αυτό είναι το μάθημα που έμαθα και που διδάσκω στους φοιτητές μου συνήθως ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς ως βουλευτές του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αυτής γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να είναι προσβάσιμη η δημόσια διοίκηση και η πείρα μου στο θέμα αυτό φαίνεται από το βιογραφικό μου σημείωμα. Και το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα μπροστά σας σημαίνει ότι θεωρήσατε παραδεκτή την υποψηφιότητά μου. Για οποιασδήποτε άλλες διευκρινήσεις βρίσκομαι στη διάθεσή σας. Επιπλέον, Ήδη έχω απαντήσει γραπτός κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για σχετικά ζητήματα. Οι απαντήσεις μου αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες μου όσον αφορά τις υπηρεσίες του διαμεσολαβητή. Και για να έχει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα. Υπάρχει όμως μια βασική αρχή μια θεμελιώδης αρχή την οποία θα πρέπει να επαναλάβω. Η επίσημη αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνεται στα συντάγματα όλων των κρατών μελών δεν αρκεί για να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Η προστασία των δικαιωμάτων αυτών Και μιλάω για την προστασία που παρέχει ο διαμεσολαβητής. Η προστασία αυτή δεν είναι η ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλες τις περιφέρειες. Και υπάρχουν σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα και από περιφέρεια σε περιφέρεια. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης ε, που έγινε στη Φλωρεντία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του φορέα αυτού, ε, είδαμε το εξής αποτέλεσμα, ότι σε πολλά κράτη-μέλη και σε πολλές περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταργηθεί δια νόμου ο διαμεσολαβητής ή ο συνήγορος του πολίτη. Άλλοι δεν επαναδιορίστηκαν και άλλοι συνήγοροι του πολίτη έχουν αποκτήσει μικρότερη αξία, έχουν υποβαθμιστεί. Αυτά είναι γνωστά εδώ και καιρό και υπό το φως αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Καταρχήν, ποιες είναι οι αιτίες της αρνητικής αυτής τάσης. Δεύτερον, τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για το θέμα αυτό. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, οι λόγοι είναι σαφείς σε οποιονδήποτε ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει καθημερινές επαφές με τη δημόσια διοίκηση. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι το Κοινοβούλιο και η τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι δομές που έχουν καθιερωθεί για να υπάρχει διοίκηση μιας χώρας και για να υπάρχει ευημερία σε μια χώρα αυτή. Κάποια στιγμή όμως οι φορείς αυτοί ε, μπορεί να γίνουν σκοπός να αποκτήσουν δική τους κυριαρχία και μάλιστα όχι μέσα στο συγκεκριμένο περιορισμένο χώρο τους, αλλά με αξιώσεις για οικουμενικότητα. Τα... Οι φορείς αυτοί λοιπόν δεν προστατεύουν πάντα τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι γίνονται μέσω για τις ε, αρχές και έτσι οι αρχές αυτές δεν πληρούν πια τον ρόλο τους να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι σαφές ότι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να υφίστανται διακρίσεις, διότι έχουν κοινή την ίδια υπηκότητα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία τους και για όλους τους συνηγόρους του πολίτη που συνδέονται μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου να έχουν ένα σαφέ ευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Σε περιπτώσεις λοιπόν σαφών διακρίσεων, θα πετύχουμε με αποτελεσματικότητα εάν κατόπιν συμφωνίας με το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την Επιτροπή σας βρεθεί μια λύση. Γνωρίζω ότι μετά από 10 χρόνια αφοσίωσης στους πολίτες της χώρας μου και της περιφέρειάς μου, η δέσμευση να παράσχω καλές υπηρεσίες είναι ακόμα πιο δυνατή. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Honorable President. Κυρία Πρόεδρε, ολοκλήρωσα την εισαγωγή μου. Νομίζω όμως ότι πολλές άλλες σημαντικές πτυχές μπορούν να αναλυθούν με περισσότερες λεπτομέρειες και θα προκύψουν από τις ερωτήσεις σας. Κυρία Πρόεδρε, Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα από το και Εξαιτία Εξαιτίας της φύση αυτή τη φύσης αυτής έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Για να είμαι σίγουρος λοιπόν ότι εκφράζομαι σωστά, θα εκφραστώ στη μητρική μου γλώσσα στη συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Βιτόριο Μπότολη για την εισήγηση αυτή. Βεβαίως ε, θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε και να τον συγχαρούμε. Έχουν οι συνάδελφοι το λόγο και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που σας έχουμε δώσει, ο καθένας μπορεί να παρέμβει δύο λεπτά. Η κυρία Γκρουνή είναι η πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Μπότολη. Οι ερωτήσεις μου. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του επόμενου διαμεσολαβητή, για την επόμενη δηλαδή θητεία, αρχές ε, οι βελτιώσεις του ρόλου αυτού και κατά πόσο θα αλλάξει το οργανόγραμμα. Τι προβλέπουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να βελτιώσουν αυτή την υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των πολιτών και το ρόλο του Ombudsman όπως ορίζεται στις συνθήκες. Ποια είναι τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο θεσμών και θεσμικών οργάνων, πώς ε, προβλέπετε την συνεργασία σας με την Επιτροπή Αναφορών, καθώς και με, τους, με τα άλλα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Γκρουνή. Ο κύριος Μποσινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε με καθηγητά. Να σας ρωτήσω το εξής. Τι προτείνετε για να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού, μάλλον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των εθνικών ομολόγων του σε εθνικό επίπεδο.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 Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα δικαιώματα των ε, εθνοτικών μειονοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Αυτά τα δικαιώματα φαίνεται να έχουν περιθωριοποιηθεί και ίσως η αιτία είναι ότι δεν θέλουμε να πλεχτούμε σε διάφορες συγκρούσεις που προκύπτουν από τα προβλήματα αυτά. Πολλοί ωστόσο πιστεύουν ότι τέτοιες συγκρούσεις θα μπορούσαν να επιληθούν μέσω του διαλόγου. Δεν είναι καλή ιδέα να υποκρινόμαστε ότι αυτά τα προβλήματα, αυτές οι συγκρούσεις δεν υφίστανται. Ίσως λοιπόν ο διαμεσολαβητής θα μπορούσε να βοηθήσει, να συνδράμει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξή. Και θα τη θέσω την ερώτηση αυτή και στους άλλους δύο υποψηφίους τα δικαιώματα των μειονοτήτων μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στο μέλλον θα τύχουν τις ίδιες αντιμετώπισης και ότι θα αντιμετωπιστούν ως συγκεκριμένο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, περιπτώσεις παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και άλλων τέτοιων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό αυτό γιατί πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουγγαρία μεταξύ αυτών Πολλοί άνθρωποι λοιπόν στις χώρες αυτές έχουν την αίσθηση ότι τα δικαιώματα αυτά καταπατούνται και μάλιστα αγανακτούν γιατί δεν έχουν την αίσθηση ότι δίνεται προσοχή σε αυτή την παραβίαση των δικαιωμάτων. Ρωτάω λοιπόν το εξή. Συχνά οι εθνικές πολιτικές στρέφονται κατά των δικών μας πολιτικών, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κοινέ δεδηλωμένε αξίε, οι οποίε εκφράζονται μέσω πολιτικών συγκεκριμένων. Τι γίνεται, έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Έχετε συγκεκριμένα σχέδια για την ευθυγράμμιση των εθνικών πολιτικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών, προκειμένου να μην έχουν οι πολίτες την αίσθηση ότι όντως υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε ό,τι αφορά την παραβίαση του δικαιώματος έκφρασης στην Ιταλία και τελικά αν θα αποφασιστεί ότι υπήρξε τέτοια παραβίαση, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες παραβιάσεις που αφορούν τεράστιες ομάδες του πληθυσμού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ρωτήσω ποια είναι η στάση σας έναντι των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η στάση σας, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών σε ό,τι αφορά τις εθνικά δικαιώματα των μειονοτήτων. Ε, να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ε, ότι βρίσκεται μαζί μας. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση κύριε Μπότολη. Ε, ποιο ήταν το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ως εθνικός διαμεσολαβητής και ε, με ποιον τρόπο προσπαθήσατε να το λύσετε και αν εκτιμάτε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και στην Ευρώπη ή τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε είναι εντελώ διαφορετικά ως Ευρωπαίος διαμεσολαβητής. Ευχαριστώ. Grazie, Thank you, Madam Chair. And... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μπότολη στην σημερινή μας συνεδρία. Συζητώ συγγνώμη που δεν άκουσα όλη την παρουσίαση σας, άκουσα όμως το μεγαλύτερο μέρος. Τέσσερις ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. Καταρχήν κύριε Μπότολη, ο κανονισμός περί διαφάνειας 1049 αναφέρεται στις διοικητικέ δραστηριότητες των θεσμικών οργάτων καθώς και στα κράτη-μέλη, καθώς και στην εφαρμογή του ε, κοινοτικού νόμου. Υπάρχουν κανόνες σε ευρωπαϊκό και επίπεδο και σε κρατικό επίπεδο που διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς πώς θα διασφαλίσετε τα δικαιώματα που ε, θεσπίζονται εκεί να προστατευτούν, ε, να μπορούν να εφαρμοστούν δηλαδή από τους πολίτες. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι πολύ πιο σύντομη. Εσείς προσωπικά πώς θα συμβάλλετε στη βελτίωση της ε, νοοτροπίας της υπηρεσίας, ε, των, του, ε, της υπηρεσίας σας. Και τέλος, όσον αφορά αυτό που είπατε για το ότι οι υπηρεσίες γίνονται αυτοσκοπός ε, αντί να εξυπηρετούν το πολίτη, εσείς πώς θα διασφαλίσετε ο φορέας του διαμεσολαβητή να μην ε, καταλήξει έτσι και τέλος. Επειδή ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, συνήθως έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι θεσμός φιλικός προς, προς τον πολίτη, ιδιαίτερα υπό το φως ότι οι πολίτες συχνά δεν ξέρουν ε, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ένα θεσμικό όργανο και στο άλλο. Πολλοί από εμά ε, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν συνειδητοποιούμε ότι ο πολίτης δεν γνωρίζει πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ να σας ευχαριστήσω και εγώ που ήρθατε. Θα επικεντρωθώ σε μία ερώτηση που βρίσκω ότι είναι ζωτική σημασία για τον διαμεσολαβητή. Το θέμα της καλής διακυβέρνησης και των καλών πρακτικών. Τις οποίες θα πρέπει να εξετάζει ο διαμεσολαβητή πολίτη στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχετε τη νομική βάση δύο νέα άρθρα σύμφωνα με τα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την καλή διακυβέρνηση σε όλα τα θεσμικά όργανα. Εσείς πώς θα εφαρμόσετε αυτά τα άρθρα για να ισχύουν οι κανόνες αυτοί για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σαλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Μποτολή που τιμάτε με την παρουσία σας στη συνεδρίασή μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Έχω την εντύπωση και την εντύπωση αυτή την έχουν και πολλοί ότι αλλάζουν πολλά πράγματα και με μεγάλες ταχύτητες στην εποχή μας και ιδιαίτερα στην Ευρώπη λόγω της μετανάστευσης, της ε, εμφυλοχωρήσεως ατόμων με διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική θρησκεία, διαφορετικές, διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της ζωής. Ήδη πρόσφατα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επί θέματος που αφορά την Ιταλική κυβέρνηση και την Ιταλική πολιτεία έκρινε το θέμα του Σταυρού ότι είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο πρέπει να προχωρήσει στην ε, απομάκρυνση του Σταυρού από τα σχολεία, πράγμα το οποίο από τη μία πλευρά θίγει την πεποίθηση των αυτοχθόνων Ιταλών, οι οποίοι όπως ξέρουμε είναι καθολικοί χριστιανοί, και από την άλλη η διατήρησή του θίγει τους μετανάστες άλλης αυτό και μόνο το παράδειγμα δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διασφάλιση στην ισορροπία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς το ρόλο του Ευρωπαίου Μεσολαβητή στη διασφάλιση της ισορροπίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποια είναι τα όρια κατά την αποψή σας στη σύγκρουση των αγαθών και των αξιών τα οποία προανέφερα και τα οποία κατ' επέκταση είναι και πολλά άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τελειώσαμε με τις ε, προγραμματισμένες παρεμβάσεις. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Βιτόριο Μπότολη για να απαντήσει και στη συνέχεια μετά τον πρώτο γύρο θα έχετε χρόνο μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Eye. Ο κύριος Μπότολη έχει το λόγο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσω να απαντήσω πλήρως όσο το δυνατόν πληρέστερα σε αυτές τις ερωτήσεις σε σχέση με τον ρόλο του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή ιδιαίτερα πέρα από το θεσμό του Ομπούτσμαν γενικότερα. Βελτιώσεις ποιες βελτιώσεις θα ήθελε να εισαγάγει ο υποφαινόμενος εάν εκλεγεί ε, αύριο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Έχω ήδη δώσει απάντηση γραπτό στις γραπτές ερωτήσεις που μου έχει υποβάλει η Επιτροπή σας. Θα πρέπει όμως να επαναλάβω αυτή την έννοια. Πιστεύουμε ότι σημαντικό δεν είναι μόνο να τονίσουμε το εύρος της δραστηριότητας και τα θεμέλια δημιουργίας αυτού του θεσμού σε όλες τις χώρες και σε όλες τις περιφέρειες, δηλαδή η αρρωγή προς τον πολίτη ως προς τις σχέσεις του με τη δημόσια διοίκηση. Όταν ο πολίτης θεωρεί ότι κάποιο δικαίωμά του έχει παραβιαστεί από τη δημόσια διοίκηση. Δεν θα ήθελα να υπάρχουν αμφισημίες εδώ. Αυτό είναι και ο βασικός ρόλος του κάθε ombudsman σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια. Αλλά για τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή νομίζω ότι υπάρχει μία άλλη εξίσου σημαντική πτυχή που μέχρι σήμερα δεν έχει τονιστεί επαρκώς αναφέρομαι στο άρθρο 5 του οργανογράμματος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, όπου αναφέρεται ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργαστεί με τους συναδέλφους και με τα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα. Η συνεργασία αυτή για μένα θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω. θα πρέπει να υπάρχει ένας πιο ενεργός ρόλος του διαμεσολαβητή σε σχέση με τους άλλους ομπούτσμεν και τους θεσμούς που ασχολούνται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπα στην ε, εισήγησή μου, υπάρχουν περιφέρειες που βρίσκονται σε χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός διανόμου και για δεκάδες χρόνια οι διαμεσολαβητές δεν έχουν ε, ανανεωθεί, ας το πούμε έτσι. Δεν έχουν επανεκλεγεί. Και πολύ συχνά δεν μπορεί να γίνει πραγματική διαμεσολάβηση, δηλαδή ο Ombudsman περιορίζεται σε μία ταπέλα που υπάρχει σε ένα γραφείο. Άρα, τι εννοώ όταν λέω ότι ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής θα πρέπει να προωθήσει πολύ περισσότερο αυτή τη συνεργασία. Τη στιγμή που ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο όλων των ombudsmen σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν λέω καθημερινά, αλλά εν πάση υπάρχει μία ανταλλαγή πληροφοριών και επαφές. Όλοι γνωρίζουν αυτή την κατάσταση της αποδυνάμωσης του θεσμού του Ombudsman σε επίπεδο ορισμένων κρατών ή κράτους γενικότερα. Εκεί λοιπόν που ο Ombudsman βλέπει ότι υπάρχει πρόδειλη παραβίαση δικαιωμάτων του πολίτη, θα πρέπει να υπάρχει μία όχι μόνο ε, δικαιοδοτική εποπτεία, αλλά και μη δικαιοδοτική, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ κρατών και μεταξύ περιφερειών, κάτι το οποίο επισυμβαίνει σήμερα. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής. που έρχεται σε επαφή με το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την Επιτροπή Αναφορών να καταγγέλει αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει δια την πανοκρουσίας. Θα πρέπει όμως αυτοδικαίως ο Ομπούτσμαν να μπορέσει να αντιδράσει και μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Αναφορών. Τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι επικρίσεις, από όπου και αν προέρχονται, έτσι ώστε η Επιτροπή Αναφορών να μπορέσει να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, στη λύτευση, ας πούμε. Ως προς τα δικαίωμα των μειονοτήτων. Μία από τις βασικές δραστηριότητες του Ombudsman στα πλαίσια της προστασίας των πολιτών δεν αφορά γενικά την ε, προστασία υπό την αφαιρετική έννοια. Αλλά τα δικαιώματα δεύτερης γενεάς, όπως έλεγε ο φιλόσοφος Μπόμπιο, δηλαδή τα ε, δικαιώματα της γυναίκας, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα των μειονοτήτων, διότι αυτές είναι οι πλέον ευάλωτες κατηγορίες που χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία, διότι η προστασία του πολίτη θα πρέπει να ευαισθητοποιείται προς αυτές τις ε, κατηγορίες. Δηλαδή προς τους πιο αδύναμους και ευάλωτους της κοινωνίας μας. Όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, γνωρίζετε ότι ορισμένα κράτη έχουν ε, θεσμοθετήσει τον ομπούτσμαν, ο οποίος έχει αυτή την εξειδίκευση, δηλαδή την ε, υποστήριξη των μειονοτήτων. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε ομπούτσμαν θα πρέπει να προστατεύει τους πλέον ευάλωτους, τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες. Ποιο είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Ombudsman δηλαδή στα 10 χρόνια δραστηριότητάς μου στην Επιτροπή του Βένετο σε σχέση με αρμοδιότητες που αφορούν ολόκληρη τη χώρα, δηλαδή την Ιταλία, διότι θα γνωρίζετε ότι στην Ιταλία ε, δεν υπάρχει ο θεσμός του εθνικού ομπούτσμαν. Εδώ και 50 χρόνια περιμένουμε ένα τέτοιο διορισμό. Υπάρχει λοιπόν περιφερειακός ομπούτσμαν, ο οποίος έχει αρμοδιότητες και στα πλαίσια του κεντρικού κράτους. Ποιο είναι το πιο μείζον πρόβλημα που αντιμετώπισε αυτή τη δεκαετία. Η απομόνωση. Η απομόνωση της περιφέρειας του Βένετο γιατί εμείς θέλαμε να προωθήσουμε αυτή τη δραστηριότητα. Από τις ε, αιτήσει το 2001 περάσαμε στις 11.000 πέρσι, που πιστοποιούνται από μία εποπτική αρχή. Και αυτό επειδή πέρα από τη βασική δραστηριότητα του Ombudsman προώθησα και μία επικοινωνιακή δραστηριότητα, διότι κανένα στην περιφέρεια, μιλώ για τους πολίτες της περιφέρειας, κανείς δεν γνώρισε ότι υπάρχει αυτός ο θεσμός. Υπάρχει αυτό το πρόσωπο που ασχολείται με τους πολίτες. Άρα ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προωθήσει ε, το πολιτισμικό υπόβαθρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό θα πρέπει να γίνει και από τους ακαδημαϊκούς κύκλους μέσω συναντήσεων, μέσω επαφών που υπάρχουν με όλες, όλους τους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα που άπτονται του προβλήματος, αλλά επίσης θα πρέπει να ασχολείται και η περιφέρεια εκεί όπου υπάρχει αυτός ο θεσμός ο οποίος μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών τη στιγμή που υπάρχει παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων από την ε, δημόσια διοίκηση. Μίλησα για απομόνωση και απομονωτισμό. Στην περιφέρεια του Βένετο δεν υπάρχει μία επιτροπή, επιτροπή αναφορών. Άρα υπάρχει ένας μονοκρατισμός. Δηλαδή, θέλουμε βεβαίως να δώσουμε να υπάρχει μια ορατότητα, ένας ορίζοντας, έτσι ώστε να προωθούνται συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, αλλά αυτό που έχει σημασία για κάθε ombudsman είναι να έχει σημεία αναφοράς, όπως ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ε, τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το εφαλτήριο της Επιτροπής Αναφορών. Γι' αυτό προσπάθησα χρόνο με το χρόνο να δημιουργήσω μία τέτοια επιτροπή η οποία πλαισιώνεται από δημοτικούς συμβούλους ή περιφερειακούς συμβούλους που είχαν ευαισθητοποιηθεί σε αυτό το θέμα της εποπτείας και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών οι οποίοι με βοηθούσαν όχι μόνο να μην ε, θεωρήσω αυτόν απομονωμένο, αλλά με υποστήριξαν και σε όλες τις πρωτοβουλίες που έκρινα αναγκαίες για την ε, προστασία του πολίτη. Μου υποβλήθηκε και μία άλλη ερώτηση σε σχέση με την προσπελασιμότητα στην πληροφόρηση και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν. Η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα είναι ο βασικός νόμος, ο θεμελιώδης νόμος κάθε κράτους και κάθε περιφέρειας για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτός είναι ο θεμελιώδης κανόνας. Γι' αυτό, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όλα τα κράτη-μέλη μελέτησαν το θέμα και έθεσαν, έθεσαν επιτάπητος το θέμα της πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και αρχεία. Είμαι λοιπόν ικανοποιημένος από τον νόμο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως γνωρίζετε, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της δημόσιας διοίκησης. Βεβαίως ε, δεν γίνεται κατάχρηση και σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, αλλά έχει δικαίωμα πρόσβαση σε όλα τα δημόσια έγγραφα. Άρα όλοι οι πολίτες ξέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, διότι μέσω του Ombudsman οποιοδήποτε πολίτης έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Αν και την επαύριο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, δεν μπορούν να κοινοποιηθούν ούτε καν στον άμεσα ενδιαφερόμενο. Μπορεί όμως να μεσολαβήσει για να προασπίσει τα συμφέροντα του πολίτη και μέσα στα πλαίσια εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μειώσουμε και να συρρυκνώσουμε αυτή την ιερά αρχή της προσπελασιμότητας στα έγγραφα της δημόσιας διοίκησης. Ως προς τους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα. που αυτοβούλως δρούν. Αυτό είναι και το θεμελιώδες ζήτημα της δραστηριότητας του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Όλα τα συντάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανθρωποκεντρικά. Άρα το φυσικό πρόσωπο, τα φυσικά πρόσωπα είναι η πραγματική κυρίαρχη. Η δημόσια διοίκηση στην ουσία υποστηρίζει αυτή την κυριαρχία του πολίτη και την υπηρετεί. Αλλά εάν αυτό το όργανο που υπηρετεί τον πολίτη λησμονεί ότι αυτή είναι η βασική του δραστηριότητα και υποχρέωση, τότε αυτό βούλος θα πρέπει ο πολίτης να τον επαναφέρει στην τάξη. Δηλαδή, η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον πολίτη. Αυτό ορίζεται από όλα τα συντάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει οι δημόσιες διοικήσεις να ξεχνάνε τον πρωταρχικό τους ρόλο και να χρησιμοποιούν τους πολίτες μόνο όταν θα πρέπει οι πολίτες να εκλέξουν τους εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης. Αυτό είναι ύψης της σημασίας για μας. Και δυστυχώς τα παραδείγματα που σας, έδειξα, που σας έδωσα πριν καταδεικνύουν ότι ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφίστανται αυτά τα προβλήματα, διότι όταν σε μια Ιταλική περιφέρεια 20 χρόνια μετά από την δημιουργία του περιφερειακού ομπούτσμαν Όταν ένας νόμος κατάργησε αυτόν τον ομπουτσμαν μέσα σε 20 λεπτά και άρα γίνονται διακρίσεις εις βάρος αυτής της περιφέρειας σε σχέση με άλλες περιφέρειες της ίδιας της χώρας, αναρωτιέμαι κατά πόσο οι πολιτικοί που ψήφισαν αυτό τον νόμο δεν ξέχασαν ότι αφαίρεσαν από τον πληθυσμό αυτό την δυνατότητα προστασίας των συμφερόντων του. Διότι αυτό είναι το βασικότερο σημείο. Δηλαδή, όχι μόνο να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα, αλλά να τα προστατεύσουμε. Και η προστασία μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοτικής δραστηριότητας ή της εξοδικαστικής δραστηριότητας του Ombudsman. Αλλά σήμερα σε αυτή τη στιγμή που ζούμε μια μεγάλη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ποιοι είναι οι πολίτες οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν όταν παραβιάζεται ένα δικαίωμά τους, πώς μπορούν να υποστηρίξουν μία δράση και να προβούν σε μία προσφυγή. Τη στιγμή πρόκειται για μία δαπανηρή διαδικασία. Και αυτό δεν αφορά μόνο την ε, περιφέρεια του Βένετο, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλάμε για μια βραδιπορία. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Ombudsman μπορεί να δράσει με σπουδή και ανεξάρτητα, διότι δεν δεσμεύεται από ε, διοικητικές, ε, διοικητικής μορφής περιορισμού περιορισμούς. Υπάρχει μια φιλική σχέση δηλαδή έτσι ώστε να επιληθούν φιλικά και τα προβλήματα του πολίτη. Εξοδικαστικά. Και εάν δεν επιληθούν, τότε ο Ομπούτσμαν οφείλει να παρεμβεί. Όχι φιλικά, αλλά με σπουδή και με την αυστηρότητα που επιβάλλεται. Τέλος, νομίζω ότι μια άλλη σημαντική πτυχή που επαναλαμβάνω είναι η πτυχή της επικοινωνίας και ιδιαίτερα ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της Ευρώπης, όχι μόνο τα κοινοβούλια, όχι μόνο οι πολιτικοί, αλλά οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωρίζουν αυτό το θεσμό και στις σχέσεις τους με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ξέρουν ότι έχουν έναν Ευρωπαίο Ομπούτσμαν που θα τους υπερασπιστεί πάντα. Αυτός ο θεσμός δεν είναι γνωστός σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης. Τον γνωρίζουν βεβαίως οι μικρές κοινωνίες και κοινότητας. Στην Ευρώπη είναι δύσκολο κάτι τέτοιο, διότι ο Ευρωπαίος ε, διαμεσολαβητής είναι μακριά από τα κράτη-μέλη, από τις πόλεις. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής να γίνει γνωστό σε όλα τα επίπεδα. Έφερα εδώ μαζί μου και ελπίζω να μην θεωρείτε ότι σας ε, δωροδοκώ ή σας διαφύρω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών. Είναι η τελευταία εργασία του δικού μου γραφείου. Είναι ένα, ε, όπως βλέπετε, ένα στην ουσία βιβλίο υπό μορφή κόμιξ. Σε 15 λεπτά ένα παιδί της μέσης εκπαίδευσης είναι σε θέση να γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα θεμελιώδη του δικαιώματα. Υπάρχει το δικαίωμα της οικογένειας, το, τα εργασιακά δικαιώματα, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και το καθεξής. Δηλαδή, ξεκινώντας από τον πρώτο ομπούτσμαν της ιστορίας. Η Ρώμη έγινε ρες publica, δηλαδή θέμα όλων, υπόθεση όλων, διότι ο λαός επανήλθε στη Ρώμη όταν απέκτησε τον δικό του ομπούτσμαν μέσα στα πλαίσια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει γνωστοποίηση του ρόλου του ομπούτσμαν. Με συγχωρείτε εάν ε, δεν απάντησα σε όλα τα ερωτήματα, αλλά όταν μιλάει κανείς ε, ελεύθερα, ίσως καμιά φορά ε, παραβλέπει ορισμένες πτυχές. Αν ναι, να μου τις υπενθυμίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και θα ήθελα να σας χαιρετήσω. Ο κύριος Γκόμες ζήτησε το λόγο όμως τώρα μέσα στα πλαίσια του Catch Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπότολη. Εν μέρει απαντήσατε ήδη στο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Θα ήθελα όμως να το πάω και λίγο παραπέρα. Είναι πολύ εντυπωσιακή η μέθοδό σας να διαφημίζετε τις δραστηριότητές σας ε, και τις ε, δραστηριότητες στα μαθήματά σας. Το, στην περιφέρεια του Βενέτο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά για το διαμεσολαβητή. Πώς θα επιλέξετε να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο σε ό,τι αφορά την θέση, τον θεσμό αυτό. Ευχαριστώ. Κέλνερ. Thank Um, Ευχαριστώ να θέσω μία ερώτηση γιατί εξηγήσατε πώς βλέπετε το ρόλο σας έναντι των εθνικών συνηγόρων και διαμεσολαβητών και των πολιτών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η σχέση σας με τις άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες όπως Europol, με την Τράπεζα Επενδύσεων Όλοι αυτοί οι θεσμοί σχετίζονται με τον πολίτη, αναφέρονται στον πολίτη. Πώς θέλετε λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ο ρόλο του διαμεσολαβητή σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές. Äh, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μπότολη, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Να ζητήσω συγγνώμη που έχασα την εισαγωγική σας ε, παρέμβαση. Ε, μια συμπληρωματική ερώτηση όμως που ταιριάζει πολύ με αυτή που μόλις ακούσαμε. Έχουμε την Επιτροπή Αναφορών, έχουμε τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή, είναι και οι δύο φορείς που αποτελούν ένα σεισμογράφο για την Ευρώπη. Όταν πάει καλά η Ευρώπη δεν ε, λαμβάνουμε πολλές αναφορές, ενώ αντιστρόφως όταν δεν πάει καλά η Ευρώπη λαμβάνουμε πολλές. Εσείς είπατε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει κατανοητή και αποδεχτού από τους πολίτες. Εμένα με ενδιαφέρει Πώς φαντάζεστε τη συνεργασία ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Μεσολαβητή και την Επιτροπή Αναφορών. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, πώς μπορούμε να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη συνεργασία αυτή και η δεύτερη ερώτηση, Πιο ωραίε είναι οι αναφορέ όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τις, τους πολίτες. Μπορεί να μην μας ευχαριστούν οι πολίτες μετά, αλλά νιώθουμε την ε, προσωπική ικανοποίηση. Λαμβάνουμε όμως και αναφορές όπου νιώθουμε ότι θα, θα, θα θέλαμε να βοηθήσουμε. Αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν παραθυράκια, κάποια κενά σε οδηγίες και κανονισμούς. Θα μπορούσατε να φανταστείτε μια κατάσταση όπου να επισημαίνετε στο Κοινοβούλιο ότι εδώ υπάρχουν κάποια κενά στην νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ίσως θέλετε ε, μια διευκρίνηση γιατί έχετε ήδη παρέμβει. Ε, επειδή δεν μου απαντήθηκε το ερώτημά μου σχετικά με τα όρια τα οποία α, τάσσονται στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και επειδή πιστεύω ότι η αποτελεσματικότητα ενός θεσμού έχει σημασία και όχι η ρομαντική περιγραφή του θεσμού. Θα ήθελα να έχω την άποψη του κυρίου Βότολη πάνω στο θέμα του ποια είναι η άποψή του και πώς βλέπει το ρόλο του Ευρωπαίου Μεσολαβητή στη διασφάλιση της ισορροπίας αυτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποια τα όρια στη σύγκρουση καθηκόντων και στη σύγκρουση αγαθών και αξιών η οποία παρουσιάζεται στις μέρες μας όλο και πιο έντονη. Εάν δούμε τη ρομαντική άποψη του θέματος, φτιάχνουμε ένα θεσμό ο οποίος είναι απογυμνωμένος. Εγώ πιστεύω ότι ο Όμπουσμαν πρέπει να γίνει ουσιαστικός θεσμός, διότι η δικαιοσύνη αργεί. Ο Όμπουσμαν σαν εξοδικαστική λύση προβλημάτων, ιδιαίτερα στα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει και ταχύτητα να έχει και αποτελεσματικότητα και ρεαλισμό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου προσδιορίσετε κατά την άποψή σα τα όρια των καθη... της συγκρούσεως καθηκόντων τα οποία ως ημέρα έρχονται στο φως της πραγματικότητας της ευρωπαϊκής. Να σας ε, ρωτήσω το εξής για να αποφύγουμε τις παρανοήσεις γιατί είτε η Επιτροπή, μάλλον και η Επιτροπή μας και ο Διαμεσολαβητής, ε, δεν είμαστε ο Άγιος Βασίλης. Είναι σημαντικό να περιοριστούμε στις αρμοδιότητες μας. Να παραμείνουμε στο πεδίο αρμοδιότητων του διαμεσολαβητή. Μπορούμε να μιλάμε για δικαιώματα των μειονοτήτων, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από όσο ξέρω όμως δεν έχει αρμοδιότητες ο διαμεσολαβητής σε αυτά τα πεδία. Σας παρακαλώ λοιπόν να λάβετε υπόψη ότι είναι καλά ορισμένε αυτέ οι αρμοδιότητε και θα πρέπει σε αυτέ να αναφερόμαστε, στι αρμοδιότητε δηλαδή του διαμεσολαβητή. Σωστό κύριε Μποσινάρου, διότι αυτές οι αξιολογήσεις ε, αφορούν πολιτικές πτυχές που δεν σχετίζονται με, με το λειτουργήμα του διαμεσολαβητή. Εγώ εξαιτίας του ρόλου μου θα ήθελα να ζητήσω στον κύριο Μπότολη να απαντήσει, έχει το λόγο για ακόμα 7 λεπτά και να μας πει συγκεκριμένα πώς θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Αναφορών. Ποιες, ποιοι είναι οι μηχανισμοί, ενδεχόμενοι μηχανισμοί, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι πιο παραγωγική και η Επιτροπή Αναφορών αλλά και ο θεσμός του Ombudsman για να προασπίσουν την προστασία, την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη. Έχει το λόγο κύριε Μπότολη. Νομίζω ότι μίλησα για τον, ως προς το επικοινωνιακό σκέλος τα θεσμικά όργανα πολλαπλασιάζονται. Υπάρχει αυτός ο πολλαπλασιαστικός παράγων και τα μέσα κοινοποίηση των αλλαγών στο, στο, στους πληθυσμούς ε, αποκλίνουν. Δηλαδή ένα διαφημιστικό σποτ υπομορφή καρτούν μπορεί να είναι πιο αποδοτικό υπομορφή κινούμενων σχεδίων καθώς και μία σειρά επεισοδίων όπου ο πολίτης μπορούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικός με τον ομπούτσμαν και να υποβάλει το ερώτημά του. Διαπιστώσαμε την επομένη ότι υπήρχαν όλο ένα και περισσότερες αιτήσει στη συνέχεια μέσω σχολείων να έρθουμε σε επαφή με τους ε, επιθεωρητές εκπαίδευσης, να προωθήσουμε δελτία, να έρθουμε σε επαφή με επαγγελματικούς κλάδους. Υπάρχει πληθώρα μορφών, χρειάζεται και φαντασία. Θα πρέπει όμως να υπάρχει η βασική δέσμευση, ότι δηλαδή ο διαμεσολαβητής δεν πρέπει να περιορίζεται στη δραστηριότητά του, στη διοικητική του δραστηριότητα. Θα πρέπει να διαδίδει αυτές τις γνώσεις, γνώσεις που αφορούν και το γνωστικό του αντικείμενο. Τώρα, ως προς τη σχέση ε, με τους άλλους φορείς. Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση Όσο περισσότερο συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση, τόσο τα θεσμικά όργανα θα είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο Ombudsman διαδραματίζει ρόλο εισαγγελέα ή έχει ανακριτικό ρόλο. Τη στιγμή που η συνεργασία αυτή δείξει ότι υπάρχει πρόδειλη παραβίαση ενός δικαιώματος που δεν αναγνωρίζει η δημόσια διοίκηση, που παραβίασε το δικαίωμα του πολίτη, βεβαίως θα αλλάξει και η θέση του διαμεσολαβητή. Δεν θα είναι ο μελιστάλλακτος διαμεσολαβητής, αλλά θα παρέμβει δυναμικά για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη οι σχέσεις τώρα ως προς σχέση με την Επιτροπή Αναφορών. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Όταν σας είπα γιατί αισθάνομαι, αισθανόμουν μόνος στη δική μου περιφέρεια, γιατί δεν πλαισιωνόμουν από μια Επιτροπή Αναφορών. Αυτό, αυτό που έχει σημασία είναι η αγαστή συνεργασία με ένα τέτοιο όργανο. έχει μεγάλη σημασία ο πολλαπλασιαστικός ρόλος που μπορεί να ε, εξευρεθεί και μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Αναφορών. Γι' αυτό μιλάμε για μονοκρατισμό του Ombudsman, αλλά μέσα στα πλαίσια της ε, πλαισίου αυτής από την Επιτροπή Αναφορών υπάρχει ένας συλλογικός χαρακτήρας διοίκησης. Άρα μέγιστη δυνατή συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα, αλλά ιδιαίτερα με την Επιτροπή Αναφορών. Επίσης, στην τελευταία παρέμβαση ε, ελέγχθη ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε πολιτική χρειά στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά να μιλήσουμε για τα προνόμια και τα καθήκοντα του ομπουτσμαν. Μα ένας ε, δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την πεμπτουσία της, ε, του ρόλου του που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει μεγάλη σημασία όταν βλέπει ότι υπάρχουν διακρίσεις ή όταν γίνεται παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Εγώ, ε, εάν προστατεύω τον πολίτη και αν ο πολίτης έρθει σε μένα και μου πει ότι με ζημίωσε η δημόσια διοίκηση κατά αυτόν τον τρόπο, εγώ ακούω τον πολίτη, προσπαθώ να επιλύσω το πρόβλημά του που είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Πώς να μην ασχοληθώ με τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν όλους τους λαούς και όλες τις δημόσιες διοικήσεις. Ο συνήγορος του πολίτη είναι το κλαδί ενός μεγάλου δέντρου. Το δέντρο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεσμοί και τα θεσμικά όργανα προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κλαδί ενός γερού δέντρου και δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στον κορμό και στις ρίζες. Διαφορετικά ο Ombudsman δεν έχει λόγο ύπαρξης. Όταν λοιπόν λέω ότι διαμέσου αυτού του δικτύου θα δράσουμε, θα συνεργαστούμε και ο καθένας από μας γνωρίζει σε πραγματικά χρόνο τι συμβαίνει σε άλλα σημεία της Ευρώπης και μέσω της στενής συνεργασίας με την Επιτροπή Αναφορών, έτσι ώστε να στυλιτεύσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πολιτική χρειά σε όλα αυτά. Ο συνήγορος του πολίτη ορίζει τις περιπτώσεις και τις περιστάσεις που πρέπει να στυλιτεύσουμε. Και στη γραπτή μου απάντηση αναφέρθηκα και στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αναφορών. Θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση, συνεχής διαβούλευση, δηλαδή αν η Επιτροπή Αναφορών δεν επιτρέπει δεν επιτρέπει την παρέμβαση του Ευρωπαίου ε, Διαμεσολαβητή, δεν μπορεί να παρέμβει. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό. Γιατί συνέβη πρόσφατα σε μια περιφέρεια της χώρας μας. Ο, με συγχωρείτε, θα πρέπει να κλείνετε ο πρόεδρος, μάλλον ο Ευρωπαίος Διομεσολαβητής παρενέβη στην, ε, σε επίπεδο περιφέρειας που προήγει αυτό το νόμο, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης του νόμου, ο οποίος κατάργησε το συνήγορο του πολίτη σε αυτή την περιφέρεια της ε, Ιταλίας. Εν πάση περιπτώσει, ο οποιοδήποτε ομπούτσμαν θα πρέπει να προστατεύει κάθε περίπτωση τη στιγμή που παραβιάζονται τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε πολίτη. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Μπότολη. Σε αυτό το σημείο και ενώ θα αποχωρήσει ο κύριος Μπότολη, θα ήθελα ο κύριος Διαμαντούρος να λάβει θέση για να προχωρήσουμε με τη δεύτερη ακρόαση.